Voilà, Αγαπητοί συνάδελφοι, λέω να ξεκινήσουμε, λέει ο Πρόεδρος, γιατί έχουμε αρκετές, ε, αρκετούς καταλόγους ψηφοφορίας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός φιλανδικών, βουλγαρικών και κροατικών. Και στα Ολλανδικά μπορείτε να μιλάτε αλλά όχι να ακούτε. Λόγω ασθενεία από ό,τι φαίνεται. Θα μπορούσα να προσπαθήσω κι εγώ ίδιος, αλλά ξέρετε μεταξύ Ολλανδικών και Φλαμανδικών υπάρχουν αποχωρώσεις και δεν θα τολμούσα. Τέλος πάντων, ο κύριος ε, Κόζα δεν είναι εδώ γιατί βρίσκεται σε διεθνείς συναντήσεις σχετικά με τις αναπηρίες. Είχαμε στις 8 Νοεμβρίου έναν 7ο τριμερή διάλογο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι διαπραγματευτές ε, συνεφώνησαν για την ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη σχετικά με την προσβασιμότητα. για αγαθά και υπηρεσίες. Αυτά είναι είδη ενημέρωσης. Μπορούμε τώρα, εφόσον όλοι έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Α, πάω πολύ γρήγορα μου λένε. Συγγνώμη κυρία Χάκιν γιατί δεδομένη της διάταξης πάω γρήγορα αλλά όταν πας γρήγορα σκοντάφτης. Λοιπόν, θα δώσω για τις απαλλαγές το λόγο στην κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις ευφορίες εγκαίρως. Έξι γνωμοτήσεις, ξεκινώντας την εφαρμογή του γενικού επρολογισμού, πρώτα απ' όλα υπήρξε σημαντική βελτίωση στην συνολική εκτίμηση σφάλματος για τις καταβολές από Ευρωπαϊκή Ένωση από 4,4 το 2014% σε 2,4 το 2017. Αλλά Έχουμε ακόμα εκτιμήσεις υψηλότερων σφαλμάτων στα θέματα κοινωνικής και δαυκής συνοχής και στα θέματα απασχόλησης. Άλλο ένα σημείο που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι το ελεκτικό συνέδριο ε, έλεγξε 113 ολοκληρωμένα έργα ε, κοινωνικής και δαυκής συνοχής και το 65% εξ αυτών είχαν συστήματα μετρήσιμη αξιολόγηση με δείκτες, που σημαίνει ότι 35% δεν είχε, ε, αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να δούμε θα έλεγα, για την απαλλαγή των οργανισμών. Εκεί δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο εκτός από το ότι προχωρούμε στα εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων που είναι σημαντικό. Για τους τέσσερις οργανισμούς τους ίδιους μπορώ να σας πω ότι και για τους τέσσερις ανακοίνωσε τις συναλλαγές για το 17 το συνέδριο ότι οι συναλλαγές δηλαδή αυτές ήταν ε, νομότυπες και σωστές για, τον, ε, για το Ίδρυμα Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό ε, Ίδρυμα Εκπαίδευσης υπήρχε μια, ένα πάνελ ε, ηθικής διάστασης, αξιολόγησης ηθικής, εν το οποίο χαιρετίζουμε. Είχαμε 99,95% ποσοστό ε, υλοποίησης, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό. Για το Eurofund εξετάζουν την ε, χρησιμοποίηση λογισμικού για τους διαγωνισμούς ανάθεσης και υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τον Ιρλα... Ιρλανδικό συντελεστή ισοτιμίας σε 1,98% αν ακούσαμε καλά την ομιλήτρια και πρέπει να το δούμε αυτό. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής προσφορών και θα εγκριθεί μια πολιτική που θα προστατεύει την προστασία του ατόμου. Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες στην κομμοδότηση σχετικά. Τελευταίο σχόλιο για τους τέσσερις οργανισμούς. Τρεις εκ των τεσσάρων έχουν προχωρήσει σε πλήρης αναλύσεις για τον αντίκτυπο του Brexit, το EU Usher δεν το είχε πράξει, αλλά από ό,τι κατενόησα στο μεταξύ μάλλον έχει προχωρήσει στην αντίστοιχη εκτίμηση και αυτό. Είχα και άλλα να σας πω, αλλά αφού μας πιέζει ο χρόνος δεν θα τα πω. Ευχαριστώ την κυρία Χάρκιν. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι ακόμα. Δεν ξέρω ποιος είναι παρόν. Και, okay. Ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τον συνάδελφο Κούκαν και θα διαβάσω τη δήλωση την οποία έγραψε για αυτό το σκοπό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις ε, γνωμοδοτήσεις της. Αποτελούν μια πολύ καλή βάση εργασίας, όμως κάποια μικρά σχόλια για τους φακέλους, ε, για τα σημεία της ημερήσης διάταξης 4 σε 9. Η ομάδα μας χαιρετίζει την ε, βελτιωμένη εφαρμογή του προϋπολογισμού και παρόλο που υπάρχει μια βελτίωση, απαιτείται ακόμα ε, μεγαλύτερη βελτίωση, για παράδειγμα το περιθώριο λάθους ε, ε όσον αφορά την περιφερειακή συνοχή και την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την εργασία παραμένουν ε, πάνω από το 2% ε, του ποσοστού λάθους. Το ελεγκτικό συνέδριο δημοσίευσε ειδικέ εκθέσεις μετά το 2017 ε, που επίσης αφορούν την εφαρμογή διαφόρων πολιτικών μέσα στο 2017 όπως είναι για παράδειγμα η ειδική έκθεση για το Erasmus Plus, ε, τα εργαλεία κινητικότητας και προγράμματα ESF. Η ομάδα μου θα ε, λάβει υπόψη της κάποιες από αυτές τις συστάσεις και αντιπομονούμε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριος Γκουτιέρε για το S&D. Όχι, δεν έχουμε. ECR, η κυρία Τραπέζιους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Χάκιν το ECR λοιπόν ακολουθεί την γραμμή ότι αρχικά θα πρέπει να, δόδεις να δοθεί μια απαλλαγή εφόσον ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα το ελεγκτικό συνέδριο και στη συνέχεια ε, υπάρξει από αυτό μια ε, θετική αξιολόγηση σε περίπτωση που δεν έχει συμβεί αυτό όμως ε, με βάση τις ε, πληρωμές των τελευταίων χρόνων έχουν μειωθεί οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερος ε, για τη θετική του αξιολόγηση και ιδιαίτερος για, τα, προ, για τις πρόοδους έχουν γίνει ως τώρα. Υπάρχουν όμως μεμονωμένα σημεία τα οποία βλέπουμε κριτικά, με, με κριτικό βλέμμα ε, άλλα θέματα τα οποία υποστηρίζουμε, όπως για παράδειγμα ο γενικός προϋπολογισμός, η υπηρεσία για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας ε, και το ε, ΣΕΝΤΕΦΟΠ επίσης ε, και υπάρχουν δύο τα οποία βλέπουμε επικριτικά το Ίδρυμα για την επαγγελματική εκπαίδευση για παράδειγμα και εκεί σίγουρα θα, ε, θα υποβάλουμε σχόλια. Υπάρχουν όμως μεμονωμένα θέματα όπως για παράδειγμα η βεβαίωση για την ανεργία των νέων, η μικρόχρηματοδότηση των ε, μικρότερων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο μας απογοητεύει. Για τα διάφορα θέματα λοιπόν θα υποβάλουμε διάφορες τροπολογίες ε, και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τους πράσινους ο κύριος Μέζερικ. Υπάρχει κάποιος για τους πράσινους. Όχι, όχι για την Γκουε, ούτε το EFDD όχι. Ο κύριος Μαρτά απουσιάζει. Άρα τελειώνουμε εδώ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 6 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Θα εγκριθεί στην Επιτροπή μας 21-22 Ιανουαρίου θα ε, ψηφιστεί στην αρμόδια επιτροπή τον Φεβρουάριο 2019, την 8η-9η εβδομάδα, έγκριση στην Ολομέλεια στην δεύτερη ε, συνεδρίαση του Μαΐου, Μαρτίου 2019. Αυτά. Αν θέλετε πάρτε τις κάρτες σας και θα ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε πιο συγκεκριμένα από την γνωμοδότηση όσον αφορά το έρασμο Συμβιβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Γυρνάμε κάποιες σελίδες. 3. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο σελίδες μετά. Συμβιβαστική 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 8. Παράγραφος 1. Σημείο C. Τροπολογία 234. Τροπολογία 235. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 239. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 240. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 247. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 248. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε κάποιες σελίδες. Συμβιβαστική 9α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την συμβαστική 9α. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική 10, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 276. Υπέρ, κατά, αποχές, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη, συμβιβαστική 10. Την κάναμε, την κάναμε όμως λέει ο πρόεδρος. Όχι, 276. Με συγχωρείτε μου, 276. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Κάνουμε ηλεκτρονικό τσεκ για την 276. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 281. Υπέρ κατά αποχές επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 297. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 303. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στη συμβαστική 33. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. 21. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρι... Ε, απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 197 97 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο 99 υπέρ κατά με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43. Συμβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 με προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φτάνουμε τώρα στο εκτιμώντας 24 όπου έχουμε την 136 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Όχι. Καταπίπτει. Άρα συμβαστική 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές για να ελέγξουμε αν θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 και 151 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 152 εκτιμώντας 32 σε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε το 154 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, συμβαστική 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Εκατά. Αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 48. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 47, 171 και όχι συμβαστική όπως είπε ο πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη, ναι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 32 εγκρίνεται. Συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποιημένη έκθεση. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρασε. Με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. Περνάμε στα θεμελιώδη δικαιώματα. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική όχι, η 16 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Για τη 16 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μου ζητάνε να ελέγξω τη 17. Παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 όχι συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...34 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... 39 άρχεται η ψήφος παρακαλώ στο 39 πέρας έχει εγκριθεί λοιπόν 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 επίσης ονομαστική Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Α, να ελέγξουμε την 9. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Ενεκρίθη. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και άρα να ψηφίσουμε τώρα την έκθεση. Παρακαλώ ψηφίστε. πέρας με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνατα γυρνάμε δύο-τρει σελίδες, συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 104, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3,1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 τροπολογία 127, 128, 129, 130 και 131 δεν είναι αποδεκτά. Περνάμε στο 130 στην 132. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 134. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στο εκτιμώντας 1, 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2,1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2,2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2,3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2,4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6,1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7,1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7,2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8,1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9,1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9,2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9,3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 61. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα στο σύνολο της νομοδότησης, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Σας αφήνω να πάρετε μια μικρή ανάσα πριν περάσουμε στο τελευταίο που είναι και το πιο σημαντικό ίσως σήμερα, στην τελευταία ψηφοφορία. J'en profite pour boire un coup. Να πιούμε και κάτι περιμένοντας. Okay. Είστε έτοιμοι. Συμβεβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε κάποιες σελίδες. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. αποχέσα Εγκρίνεται. Γυρνάμε κάποιες σελίδες πάλι. Το βρήκατε. Συμβαστική 4. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάλι γυρνάμε σελίδες. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιον να μας βοηθάει, να μας αλλιώνει το δάχτυλο για να γυρνάμε τις σελίδες. Το βρήκατε όλοι. Όχι. Αγνές, το βρήκες. Όχι, το Λίπε 48 δεν είναι αποδεκτό. Ε, συμβαστική 5, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Βρήκατε όλη την συμβιβαστική 6, υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Τετρακόσια δέκα εννέα υπέρ. 419 υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 419. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 420 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση για το 420. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας για το 420. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 7 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάλι κάποιες σελίδες παρακάτω. 492. Τη βρήκατε όλοι. Άρχεται η ψηφοφορία στο 492, είναι και πάλι ονομαστική. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μαζί με την Γιούρι 78. Περνάμε στην 493 υπέρ και την Γιούρι 79 κατά συνέπεια. 493 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7α. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Γίτσες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 526. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ για το 526. Άρχεται η ψηφοφορία για την 526. Επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Και όμως... Ε, ήταν λίγο τσιματσίμα. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. «541, Ρέτζι 66 και 545 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μαζί, Ρέτζι 67 και 562, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για το Ρέτζι 67 και την 562 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 542. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Επαλήθευση για το 542. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερις σελίδες μετά. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοντ 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε κάποιες σελίδες και πάλι. Τέσσερις σελίδες μετά, συμβαστική 23α, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 69, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα. Τα άρθρα από το MV45 μέχρι το Γιούρι 65 δεν τα ψηφίζουμε γιατί είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες της MV. Περνάμε λοιπόν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 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε κάποιες σελίδες. Παράρτημα 3 από το MV78 μέχρι το 80 είναι αρμοδιότητες της MV, δεν τις ψηφίζουμε. Περνάμε λοιπόν στην αναφορά 25, εκτιμώντας 26 υπέρ κατά εγκρίνεται, συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 1 ABC νέο, φαμ 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 2 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 4 A νέο. Άρθρο 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47. Επαλήθευση για το 46. Ξανά. Με συγχωρείτε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παραλίγο. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 49, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 5, 46 Λεοπρόεδρος και Γιούρι 7. Ε, επαλήθευση 55, 56 συγγνώμη και Γιούρι 7. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Το 57, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 50, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 2, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 6, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται εκτιμώντας 8 το 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 62. Γιούρι 8 και NV4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. MV5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοντ 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 70. Όχι, καταπίπτει. Και πάμε στο 71. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 53. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ 22. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Badge 7. Τσεκ για το 82. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μπάτζ 7, επομένως, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 54, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 54α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλτ 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκτιμώντας A και b μαζί με το 98 έχουμε το Γιούρι 15 και το ΦΑΜ 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 56. Υπέρ. Κατά. Συμβεστι... Ε, αποχές. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στα εκτιμώντας 17. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι μαζί, πάει μαζί με το MV8. Κάλτ 18, όχι, καταπίπτει. 110 και Ρέτζι 13 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 10, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. NV9, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 57, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Από κοινού, 121, 122, 228 και Ρέτζι 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Να ελέγξω. 121, 122, 228 και Ρέτζι 30. Ε, ε, άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. πέρας και ενεγκρίθησαν. 58 υπέρ. Συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 100 συγγνώμη καταπίπτει Άρα από κοινού 130, όχι, από κοινού 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5. Να ελέγξουμε 130 θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ, 130. Πέρας. Απορρίπτεται οριακά. Τέλο πάντων, 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 20, 136 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε λοιπόν την 136 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 158 και αυτή και τα λοιπά. Συμβαστική 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 170 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 176, 177, 77 budget 13, κουλτ 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ε, 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 179 υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 65 υπέρ. Κατά Κατά, εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 66α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 29, 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλ 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Να ελέγξουμε λοιπόν την Κουλτ 31. Παρακαλώ. Je Πέρας. Εγκρίνεται. Λίμπε 23. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φάμ 24 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Εκτιμώντας 31. Η 204 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 205 και γιούρι 30 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνονται. Κουλ 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από ελάχιστους. Δεν βλέπω χέρια. Να ελέγξουμε λοιπόν τη 2.16 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας και απορρίπτεται λέει κατά λάθο ο πρόεδρο, ενώ εγκρίνεται, εγκρίνεται, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, περνώ στην 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κόντ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 37α λέει ο πρόεδρος εννοεί την 73α. Ναι, 73α λέει τώρα ο πρόεδρος. Σεπτών για να το πω στα βέλγικα λέει ο πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Envy 11 με λίμπε 29 είναι της ΕΝΒΗ. Περνάμε λοιπόν στην 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κόντ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπούτς 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 είπε κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε τη 229 λοιπόν παρακαλώ ψηφίστε πέρας απορρίπτεται με ίσε ψήφου. Λοιπόν, η συμβαστική 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, NV30 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Άρα τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε τελικώ για το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρα. Ιδού. tous les cas, c'était une brique. Ήταν τεράστιο το έγγραφο, αλλά συγχαρητήρια.